Ωραία. Αγαπητοί συνάδελφοι, περατώθηκε η συζήτηση. Ευχαριστούμε τον Επίτροπο, ο οποίος ε, έμεινε εδώ μέχρι το τέλος της συζήτησης. Η συνεδρίαση συνεχίζεται αύριο στις 26 Οκτωβρίου από τις 8.30 μέχρι τις 11.30 και 11.30 με 1.30. Η ημερήσια διάταξη έχει δημοσιευθεί και ε, μπορείτε να τη δείτε στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καληνύχτα σε όλους. Και